Στο τελευταίο θέμα για απόψε, παρεμβάσει διάρκεια ενό λεπτού σύμφωνα με το άρθρο 163 του κανονισμού. Το λόγο έχει ο κύριος Ξάκη για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα η πιο διαδεδομένη λέξη είναι αλληλεγγύη. Μόνο για αλληλεγγύη ακούμε. Και αλληλεγγύη είναι κάτι που επικαλείται ε, κάποιος για να αλλάξει μια ε, λάθος ε, απόφαση όπως είναι ο πολιτισμός του ευπρόσδεκτου Willkommenskultur για τους πρόσφυγες στη Γερμανία και στην Ευρώπη αλλάζει η κατάσταση, ε, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες χωρίς να το θέλουν. Σήμερα στη Σλοβακία έχουμε δασκάλους και νοσηλευτρίες που είναι στο δρόμο και διαδηλώνουν ε, για τους μισθούς και τις εργασιακές συνθήκες. Θα πρέπει να ακούμε περισσότερο τις φωνές από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Ο κόσμος υποφέρει. Ε, σας λέω, οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές ζητούν από την Ευρώπη να σταματήσουν οι εγωισμοί. Έχουμε διαρροή εγκεφάλων ε, και αυτό πλήττει σφοδρά την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ε, εμείς δεν καλύπτουμε το χάσμα με τη Δυτική Ευρώπη, χρειάζεται προσοχή γιατί κινδυνεύει η κατάσταση να εξοκέλει. Νεγκρέσκου, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο κατάρτισης της ε, πολιτικής, γιατί δεν μιλάμε για προνόμια. Η πολιτική ε, σχετίζεται με το τι θα κάνουμε για τους ανθρώπους. Θέλουμε στη Ρουμανία να καταπολεμήσουμε την φτώχεια, να προωθήσουμε την υγεία, να ε, έχουμε μία ανθρωποκεντρική πολιτική αλλά δυστυχώς ε, αύριο ποιος θα μας ακούσει. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε την οτροπία και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε και τους μηχανισμούς και τους στόχους. Οι άνθρωποι δεν έχουν πια υπομονή. Το πρώτο ε, ε, βήμα είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Στρατηγικών Επενδύσεων βοηθώντας τις ε, ΜΜΕ, έτσι ώστε να αναπτυχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιούρεκ, γιατί ο Ζωκ ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τώρα με μεγάλη προσοχή την Πολωνία, την πατρίδα μου και πολλές φορές ε, υφίσταται και επιθέσεις γιατί υποτίθεται ότι η Πολωνία παραβιάζει το άρθρο 2 λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης το, το, της συνθήκης. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ε, γιατί αυτή η κατονία. Είδατε στην κολονία τι έγινε την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ε, ε, αυτά που λέει το άρθρο 2 της συνθήκης δεν τηρούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να την πληρώνει η Πολωνία. Τι μπορούμε να πούμε. Στη Γερμανία η ε, αστυνομία κράτησε κρυφές κάποιες προφορίες από τον πληθυσμό. Η επίσημη μεταναστευτική πολιτική ε, θα κινδυνεύσει αν μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Τι σχέση έχουν όμως όλα αυτά με την Πολωνία και το δικαίωμα ε, στην ελευθερία του λόγου. Θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Τι νόημα έχουν όλες αυτές οι εξαρτήσεις. Η κυρία Μπιλμπάου Παραντίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μια χαλιβουργία στη χώρα των Βάσκων κλείνει ένα εργοστάσιο καινοτόμο της κυκλικής οικονομίας που ε, χρησιμοποιεί ε, καλές συμβάσεις για να διατηρήσει την απασχόληση. Αυτό είναι ένα σύμβολο για την ανάπτυξη 2020 και τι γίνεται με μια βιομηχανική περιοχή. Τώρα έρχεται και το ντάμπινγκ της Κίνας και η ε, κρίση στην ενεργειακή και οικονομική αγορά και κινδυνεύουν χιλιάδες οικογένειες. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτές γιατί πρώτα απ' όλα μιλάμε για ανθρώπους, για ζωή, για εφορία, για κοινωνική δικαιοσύνη είναι η ίδια η ουσία και η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιδράσουμε απέναντι ε, σε ε, ξένα προϊόντα που έρχονται με dumping. Είναι σκανδαλώδεις οι διαφορές ε, στην τιμή της ενέργειας και στην τιμή του χρήματος στην ενιαία αγορά. Πού είναι η ανταγωνιστικότητα, πού είναι η επαναβιομηχάνηση. Η κρίση ε, στη βασική χαλιβουργία είναι ένα σύμπτωμα μιας βαριάς αρρώστιας που απειλεί πολλές επιχειρήσεις, πολλές θέσεις εργασίας και χρειάζεται ε, επιγόντως να απαντήσουμε τώρα. Η πρόεδρος που απειλει πολλες επιχειρησεις πολλες θεσεις και χρειαζεται επιγοντως να απαντησουμε τωρα η προεδρος διακοπτει την ομιλήτρια. Ο κύριος Μπενίτο Σιλουάγκα. Καταρχήν, θα ήθελα να ε, δράσουμε στο, ως προς το πυρηνικό, ε, μια πυρηνική εγκατάσταση στην ε, εκλογική μου περιφέρεια, γιατί από όσο γνωρίζω θα υπήρξε μεγάλος κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς κλείνουμε τα αυτιά μας και η Στη Καρόνια και Κοφρέντες δεν γίνονται έλεγχοι των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Υπάρχουν δύο παράλληλοι αντιδραστήρες στο Βέλγιο και θα θέλαμε το ε, Συμβούλιο Πυρηνικής Ασφάλειας να λάβουν υπόψη αυτή την κατάσταση επισφάλειας. Ελπίζω να ε, μην μετατραπεί η Γκαρόνια σε μια νέα Φουκουσίμα της Ευρώπης. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Τερικάμπρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε στις 28 Οκτωβρίου λάβαμε μία απόφαση για την πρωτοβουλία των πολιτών. Δεν αντιμετωπίστηκε το θέμα ενός follow-up που θα έπρεπε να δοθεί γιατί μόνο τρεις από τις 15 προτάσεις ECI ελήφθησαν υπόψη. Δεν υπήρξε follow-up. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, αυτές οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, διότι υπάρχει ευρωσκεπτικισμός και η ίδια η Επιτροπή πλήττει τα ευρωπαϊκά αυτά σχέδια. Αυτό είναι απίστευτο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κοράου. Στην Σικελία όπως σε όλη τη Μεσόγειο η γεωργία ανθεί αν λάβουμε υπόψη τα πορτοκάλια μας, ε, τις ντομάτες και αυτό και το εξαιρετικό ελαιόλαδο που παράγουμε. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να προβάλλει αυτές, ε, αυτή την ποιότητα, την καταστρέφει διότι προέβη σε μία αύξηση συναλλαγών με το Μαρόκο και την Τινησία. Μιλά για αύξηση εισαγωγής 35.000 τόνων. Και θα ήθελα να πω τι θα γίνει Εάν δεν μπορείτε να προωθήσετε την παραγωγή, τις παραγωγές μας, αυτό σημαίνει ότι ερχόσαστε εδώ μόνο για την παρουσία σας και για τίποτα άλλο. Ρεβέκα. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Αυστρία έχει αναστείλει την, ε, το χώρο Σέγγεν. Η Ελλάδα απειλείται με αποχώρηση από το χώρο Σέγγεν. Όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο το Σέγγεν και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες και άλλοι θα ακολουθήσουν την Αυστρία. Εάν δεν το λάβετε αυτό υπόψη, η Ρουμανία μαζί με τη Βουλγαρία δεν θα μπορέσουν να προσχωρήσουν και θα πρέπει να δεχτούμε τις ευρωπαϊκές ποσοστώσεις. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δύο αυτά κράτη. Εφόσον δεν μας επιτρέπεται να προσχωρήσουμε στο χώρο Σέγγεν, τότε δεν θα μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Μπορεί να απαντήσει κανείς ε, κατά πόσο η Ρουμανία θα προσχωρήσει στο χώρο Σέγγεν. Κύριε Κόρβιν Μίκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Θέλω να μιλήσω για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται συζήτηση. Πριν από λίγα λεφτά όμως ακούσαμε εδώ μέσα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει λέει στους Κινέζους πόσο γρήγορα πρέπει να αναπτυχθούν. Και δεν γέλασε κανείς με αυτά που ακούσαμε. Οι Κινέζοι ξέρουν και αυτοί ξένες γλώσσες και ακούνε τι γίνεται εδώ μέσα και τι διαμείβεται. Και επίσης πολλές φορές είναι πολύ πιο έξυπνοι από εμά. Λοιπόν, φανταστείτε να φτάσει τα αυτιά τους αυτό που λέμε εδώ μέσα. Αν παρακολουθούν τη συζήτηση του Κοινοβουλίου, δηλαδή, θα ξεκαρδίζονται. Σας παρακαλώ λοιπόν να διατηρήσουμε ένα στοιχειώδης επίπεδο εδώ στη συζήτηση του Κοινοβουλίου. Κατά τα άλλα ξέρετε τη γνώμη μου ότι πρέπει να καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ράνς Καρσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 19 Ιανουαρίου, χωρίς προφανή λόγο ούτε ε, προειδοποίηση, η Αλτάδης ε, στη Ριόχα είπε ότι στις 30 Ιουνίου κλείνει καπνοβιομηχανία. Για ποιο λόγο, ότι η Αλτάδης ούτε είναι ελληματική η ε, επιχείρηση, 471 απολύει άμεσα και συναφείς ακόμα περισσότερους. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θα πρέπει να αποτρέψουν αυτό στην ε, περιφέρεια της Ριόχα ξεκάθαρα έχουμε πει ότι απορρίπτουμε απολύτως αυτή την αδικαιολόγητη ενέργεια, να κλείσει αυτό το εργοστάσιο και το Συμβούλιο Επιχείρησης και ο λαός της περιοχής αντιτίθεται είναι πάνω από 100 χρόνια αυτή η καπνοβιομηχανία και δημιουργεί πλούτο και θέσει απασχόληση. Και είναι σοβαρό κίνδυνο για πάνω από 10.000 οικογένειε που είναι ε, καλλιεργητέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σόνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται ότι κάποιες εκατοντάδες ε, τρομοκράτες κατάφεραν να παραλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με το φόβο. Κατάφεραν να σπείρουν το φόβο και να οδηγήσουν και σε διχόνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι καταπιέζονται τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένας τρόπος αποτελεσματικός να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Πρόκειται όμως για μία διχόνοια η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική απάντηση έναντι της τρομοκρατίας. Η Ουγγαρία και η κυβέρνησή της γνωρίζει πολύ καλά αυτό το φαινόμενο καθότι έχουμε υποβάλει μία συνταγματική μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε ακριβώς να μιλήσουμε για αυτήν την τρομοκρατική απειλή, την επιβολή για 60 μέρες της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, οι περήφανοι αγρότες της πατρίδος μου της Ελλάδος βρίσκονται στο πόδι. Βρίσκονται στα μπλόκα και πολεύουν για την ίδια τους την επιβίωση. Η Τρόικα και οι δανειστές με την μνημονιακή τους πολιτική, την οποία εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, διαλύουν το πρωτογενή τομέα επιβάλλουν φορομπηκτικό ρεσάλτο στις τσέπες των αγροτών φορολογούν άγρια τη γη που καλλιεργούν επιβάλλουν κατασχέσεις στις κοινοτικές επιδοτήσεις βάζουν χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών και διαλύουν το ασφαλιστικό του σύστημα. όμως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντιστέκονται και κλιμακώνουν το δίκαιο αγώνα τους. στο πλευρό τους βρίσκεται ολόκληρη η ελληνική κοινωνία οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι συνταξιούχοι οι εργαζόμενοι. πρόκειται για τη συγκρότηση μιας νέας κοινωνικής αντιμνημονιακής συμμαχίας που είναι αποφασισμένη να κλείσει τον δρόμο στην τρόικα μια νέα κοινωνική συμμαχία που θα εκφραστεί μαζικά δημοκρατικά και αγωνιστικά στη γενική απεργία της 4 η Φεβρουαρίου την προσεχή Πέμπτη. Γιατί όλοι οι Έλληνες παλεύουμε ενωμένοι για να πετάξουμε την Τρόικα έξω από την πατρίδα μας και να ξαναπάρουμε πίσω την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Πριν από 100 χρόνια η Ιρλανδική Δημοκρατία διακηρύχθηκε και θα πρέπει εμείς φέτος να γιορτάσουμε αυτό το γεγονός για τους αγωνιστές. Αντί να γίνει αυτό, ε, η Ιρλανδική κυβέρνηση και εδώ απέναντι κάθονται οι εκπρόσωποι της θέλουν να σβήσουν την ιστορία. Όχι μόνο ε, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. Ε, τις τελευταίες ώρες που πέρασαν οι αγωνιστές μας θέλουν να τις σβήσουν το 16. Ε, ε, σβήνουν ε, τα σημαντικότερα μουσεία, τα σημαντικότερα σημάδια. Ε, το ε, Αυτοκρατορικό Μουσείο στο Λονδίνο χαρακτήρισε την περιοχή αυτή ως την πιο άθικτη περιοχή που έγιναν εχθροπραξίες και μάχες στην Ευρώπη. Ιστορική κληρονομιά είναι και θέλουν να το κάνουν εκεί πέρα εμπορικό κέντρο και ε, θα εξυπηρετούν έτσι την αμφιλελεύθερη αζέντα τους. Θέλουν να ε, καταστρέψουν την κληρονομιά μας και αύριο θα το φέρουμε αυτό το θέμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τη η κυρία Αντινόλφη. Από όσο γνωρίζουμε, ε, έγινε, υπήρξε μία κατηγορία ε, κατά του πλουραλισμού από την κυβέρνηση μέσα στα πλαίσια των ΜΜΕ. Γιατί η Επιτροπή δεν κατηγορεί και την Ιταλική κυβέρνηση, γιατί ο Πρωθυπουργός ε, Ρέντσι μπόρεσε να διαλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρωθυπουργό της Ράισα να πρόκειτο για ένα ε, φασιστικό καθεστώς. Όπως ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση γίνεται πολιτική επιλογή και όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι εκδιώχθονται, όπως ε, ε, ισχύει στην περίπτωση του Έντσο Μπιάτζη. Τώρα τα ξέρετε όλοι. Εμείς από το κίνημα 5 αστέρων θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρεύουμε, όπως ίσχυσε και στην περίπτωση της Πολωνίας. Δεν μπορείτε Ο Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό είναι μέρο του τρίτου μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και ψήφισαν όλα τα άλλα αστικά κόμματα αποτελεί επιταγή του μεγάλου κεφαλαίου υλοποιεί στρατηγικές κατευθύνσεις ευρωπαϊκής ένωσης που προβλέπουν την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης την αντιμετώπιση της ως ατομική υπόθεση φορτώνοντας στις πλάτες των εργαζομένων αβάστακτες εισφορές μειώνοντας συντάξεις αυξάνοντας όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι τα βαθιά γεράματα η μετατροπή της σύνταξης σε επίδομα πτωχοκομείου μαζί με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας solvency ii ανοίγει το δρόμο για την αύξηση της πίτας των ομίλων ιδιωτικής ασφάλισης οι μικρομεσαίοι αγρότες επιβαρύνονται με εξοδοτικές αυξήσεις εισφορών που μαζί με τους όρους της νέας καπ τους ξεκληρίζουν πλημμυροδοτώντας τους μεγαλοαγρότες και τους ομίλους. η κυβέρνηση εδώ και τώρα να αποσύρει το νομοσχέδιο λεμιτόμο την πέμπτη στην απεργία οι εργάτες έχοντας στο πλάι τους τη μικρομεσαία αγροτιά και τα μπλόκα της τους αυταπασχολούμενους μπορούν να δώσουν μαζική αποφασιστική απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, έχει βελτιωθεί πολύ ε, η υπόθεση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και η χρηματοδότηση. Γίνεται ένας διάλογος στη Βιέννη που άρχισε την περασμένη ε, χρονιά το καλοκαίρι και ξέρουμε ότι διευρύνεται και επεκτείνεται το κεντρικό δίκτυο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και συγκεκριμένα τρία έργα είναι αυτά δύο ευρωπαϊκών δικτύων και έχουν επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. Ωραία όλα αυτά, αλλά για να μπορέσουν να ε, χρησιμοποιούνται παντού, για να ε, μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί αυτούς τους διαδρόμους χρειάζονται ε, μεταρρυθμίσεις και στον τρόπο χρηματοδότησης διότι υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα και ε, μάλιστα από υποψήφια σε υποψήφια χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί τώρα εκείνο το νομικό πλαίσιο αλλά και το οικονομικό που θα επιτρέπει τη λειτουργία αυτών των διαδρόμων. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, ευχαριστώ. Πρόκειται για σειρά προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων σε πάρα πολλούς τομείς και σε κάθε περίπτωση οι προοπτικές είναι πάρα πολύ θετικές. Χιλιάδες παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού. Στην ε, Λετωνία 23,5% των παιδιών βρίσκονται στο όριο του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Αυτά είναι τα χειρότερα νούμερα και πολλές ε, χιλιάδες παιδιών δεν μπορούν να πάνε σε σχολεία και θα πρέπει βεβαίως ε, να αλλάξει η πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά αυτό δεν αρκεί για να υπάρχει πρόσβαση στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία αυτών των παιδιών. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη στην περιοχή του Λατγκάλε όπου υπάρχει εγκατάλειψη από τους κατοίκους της περιοχής αυτής και τα προβλήματα αυτά είναι όλο και πιο σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στους πρόσφυγες και βεβαίως την άνηση κατανομή τους στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξει πολύ πιο δίκαιη κατανομή. Η Φιλανδία έχει πληγεί πολύ σημαντικά εξαιτίας των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 400 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που έχασαν οι αγρότες από την χώρα μας. Βεβαίως και δεν λέω ότι πρέπει να υπάρξει άρση των κυρώσεων γιατί θα στείλουμε λανθασμένο μήνυμα προς το Κρεμλίνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει πιο ίση και πιο δίκαιη η κατανομή του βάρους. Αυτό ισχύει για τους πρόσφυγες αλλά ισχύει και για τα αποτελέσματα των κυρώσεων. Θα πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός. Ευχαριστώ η κυρία Πάρκερ. Thank you. Ευχαριστώ. Όλοι ακούσατε την κατάσταση στην κολονία όπου γυναίκες έγιναν αντικείμενα επιθέσεων, κακομεταχείρισης και ενοχλήσεων. Πώς αφήσαμε κάτι τέτοιο να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύμβαση της Γενέβης του 1951 βεβαίως και δίνει ορισμούς για το ποιος είναι πρόσφυγας, κάποιος ο οποίος αναγκάζεται να διαφύγει από μια περιοχή από την οποία διώκεται είτε που αναγκάζεται να ξεφύγει από κακομεταχείριση λόγω της θρησκευτική ή άλλης ε, μειονότητας την οποία αρχίζει. Σε κάθε περίπτωση εδώ θα πρέπει να δούμε αν πρόκειται για άτομα που εμπίπτουν σε αυτόν τον ε, ορισμό του πρόσφυγα γιατί σε κάθε περίπτωση Αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μετανάστες, πάνω από 500.000, οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και αντιμετωπίζουν τις γυναίκες σαν πολίτες δευτέρας κατηγορίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάλεβιτς. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Οι τοπικές αρχές έχουν πολύ καλές ιδέες και προετοιμάζουν σχέδια για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών τους. Όπως για τις πράσινες μεταφορές, για την ψηφιοποίηση και ούτω καθεξής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης και η έλλειψη πληροφοριών σε σχέση με αυτά τα προγράμματα. Κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας έτσι ώστε τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα νέα επενδυτικά προγράμματα να γνωστοποιούνται εγκαίρως στις τοπικές αρχές. Δεν υπάρχει καλή διάρθρωση και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ο κύριος Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Μιλώ στην Ολοβέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταγγείλω ε, ε, την τελευταία δράση της ε, κυβέρνησης της υπηρεσιακής για το υδρολογικό σχέδιο της λεκάνης του ποταμού Εύρου της Ισπανίας και ε, ε, ε, απειλεί το δέλτα του ποταμού το οικοσύστημα και είναι και κοινωνικο-οικονομική επίθεση στην περιφέρεια. Χωρίς διάλογο έγινε αυτό με τις αρχές της Καταλωνίας, τις τοπικές. Δεν έλαβε υπόψη τη συμμετοχή των πολιτών, αγνόησε την πλατφόρμα για την ναι, υπεράσπιση του εύρου και επίσης είναι κατά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως είναι εκείνη για την προστασία των υδάτων, των οικοτόπων ή των πτηνών. Είναι σημαντικές οι κινητοποιήσεις αυτά το Σαββατοκυριακό. Ε, ε, Προσώπηση του Κοινοβουλίου θα μεταβεί στο Δέλτα του ποταμού Εύρου τη Δευτέρα και θα διεισόμαστε την κατάσταση. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, μετά από 20 χρόνια ε, μίας ε, πολιτικής δασοκομείας όπου πλούτησαν ε, οι εμπλεκόμενοι φορείς μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων επιχειρήσεων για να αγοράσουν εξοπλισμό και τρακτέρ και αφού ε, χτίσανε και δημιούργησαν επιμελητιακά κέντρα, στην ουσία ε, δεν πρόωθησαν την ε, δασοκομεία και τον δασοκομικό φορέα. Νομίζω ότι θα υπάρξουν προβλήματα στη διαχείριση της δασοκομείας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις διαφθοράς. Υπάρχουν ε, κρατικές επιδοτήσεις που υποσκάπτουν την, τον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να παρέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις και μέσα στα πλαίσια του συστήματος εκχωρήσεων θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα το δασοκομικό. Ο κύριος Γκουτιέρες δεν είναι εδώ, η κυρία Κίρτον Τάρλινγκ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις ανανεώσιμες διαφορετικά για να έχουμε ένα ε, πολύ καλύτερο ηλεκτρικό δίκτυο στη Βόρειο Θάλασσα για να έχουμε καθαρή ενέργεια και χαμηλό κόστος και να διατηρηθούν θέσεις εργασίας ε, και στην ε, εκλογική περιφέρεια στα βορειοανατολικά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Εμείς ε, προωθήσαμε ένα πρόγραμμα δράσης για την ενέργεια στη Βόρειο Θάλασσα, στην Ολλανδική Προεδρία. Αυτή την Πέμπτη θα δοθεί συνέχεια και θα ήθελα η Βόρειος Θάλασσα να γίνει μια καθαρή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για την Ευρώπη. Ο κύριος Σόγκορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οικονομική συνεργασία ε, βοηθάει για να ξεπεράσουν ε, οι χώρες τις διαφορές τους και να συμφιλειωθούν. Ε, οι ε, ιδρυτικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Γι' αυτό το λόγο ε, δημιουργήθηκαν. Στη συνέχεια οι χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν χάθηκε η δυσπιστία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες για να μην πω ε, αιώνες μεταξύ κρατών. Η καλή οικονομική συνεργασία και πολύ σημαντική αλλά χρειάζεται ειλικρινής διάλογος για τα καθόδη ζητήματα και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Εδώ αναφέρομαι κυρίως στην προστασία των ε, εθνικών μειονοτήτων. Τι θα πει αυτό το δικαίωμα δικαίωμα να έχουν την ίδια τους την ταυτότητα, την ευημερία τους, την ισότητα των δικαιωμάτων και την ύπαρξή τους στην ίδια μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν χώρες στην περιφέρεια μας, η Σλοβακία όπως η Ρουμανία, που δεν θεωρούν τις αυτόχθονες μειονότητες ως ε, αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειας, αλλά το θεωρούν απειλή και θέλουν να τους αφομοιώσουν. Και ως τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Τσεχόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, την επιμονή των Νορβηγών όσον αφορά κάποιες οικογένειες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παραδείγματος χάρη τη Σλοβακία, την Τσεχία, παραδείγματο χάρη για κάποιους παράξενους λόγους απομακρύνουν τα παιδιά από τις οικογένειές τους. Πρόκειται για μια δημοκρατική και πολιτισμένη χώρα. Και πραγματικά αυτή η κατάχρηση, αυτές οι καταχρήσεις είναι κάτι που δεν πρέπει να μας αφήσει αδιάφορους. Υπάρχουν διαδηλώσεις παντού ε, στον κόσμο και οι Ευρωπαίοι πολίτες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιτεθούν και να πούν όχι σε αυτές τις αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στις οικογενειακές τους υποθέσεις. Νομίζω ότι κύριε Επίτροπε εδώ πρέπει να αντιδράσουμε. Σαν τελευταίος ομιλητής θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχεστε και κάθεστε τόσο αργά μαζί μας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε τις ομιλίες των ΣΔΙΤΟΥ. Θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί στις 8.30 έως τις και η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευστεί στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ τους διερμηνείς που βρίσκονται εδώ